για το Γουαντάναμο που προβλεπόταν για την Πέμπτη το απόγευμα. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν θέλει τον λόγο ο κύριο Αλαφράγκα τώρα. Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα το πρωί ε, κατέθεσα αυτό το αίτημα εξ ονόματος της πολιτικής μου για να προσπαθήσουμε να σεβαστούμε τη συμφωνία της Ολομέλειας που ήταν στις 18 Απριλίου. Είχαμε αποφασίσει, θυμάστε, να συζητήσουμε τότε και να ψηφίσουμε το Μάιο. Και η Προεδρεύουσα τότε, κυρία Ποδηματά, μας είπε να το πράξουμε γραπτός. Όπερ και γένετο και είχαμε πει ότι σήμερα στις 3 το απόγευμα θα αποφασίζαμε σχετικώς. Και θα παρακαλούσα κύριε Πρόεδρε να μας διευκρινίσετε τώρα ποια ακριβώς διαδικασία ισχύει και πότε θα τελειώσουμε με αυτό το ακαθόδες ζήτημα για να μπορέσει η Ολομέλεια να ανταποκριθεί στις ευθύνες που έχει αναλάβει και όπως ε, ανέφερε το πρωί συνάδελφος Βερονίκ Τεκεζέρ εξ ονόματος της Σοσιαλιστικής Ομάδας διότι ο πρόεδρος της ομάδας ε, των Σοσιαλιστών ε, αντέταξε διαφορετική πρόταση στη δική μου και ομόφωνα η Ολομέλεια αποφάσισε. Μπορείτε κύριε Πρόεδρε τώρα να μας διαφωτίσετε. Τώρα στις 3 θα αποφασίσουμε ή μήπως θα λυθεί αυτό το θέμα αύριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. According to uh, the... Δύναμη της αποφάσεως που έχει λάβει ο πρόεδρος του σώματος θα υποβληθεί το αίτημα πριν από τη συζήτηση στην αυριανή συνεδρίαση. Δηλαδή